της τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συνεργίες μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του προγράμματο Ορίζοντα 2020 και ξεκινάει λοιπόν αυτή η συζήτηση με την δήλωση του Επιτρόπου Μοϊντά. Σα ευχαριστώ, Επιτρόπε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε για να μιλήσω στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τη σημασία των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του προγράμματο Ορίζοντα 2020. Δυστυχώ, όπω ξέρετε, η Επίτροπο Κρέτσου δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα, αλλά μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω. Παρότι οι συνέργειε συζητούνται εδώ στο Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια, ο Ορίζοντα 2020 είναι το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία που ξεκάθαρα και ρητά αναφέρεται στις συνέργειες με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και μαθητικά ταμεία. Ο κανονισμός ο οποίος ε, θέσπισε αυτά τα ταμεία ενώ στο παλιό πρόγραμμα ε, μιλούσαμε για συνέργειες που ήταν καλό να τις έχουμε, τώρα αυτό το πράγμα, οι συνέργειες έγιναν ένα απόλυτο, μια απόλυτη ε, ανάγκη, έγιναν ένα must. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω γιατί οι συνέργειες είναι τόσο θεμελιώδεις. Όσες περισσότερες έχουμε μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του ορίζοντα 2020, τόσο περισσότερη επίπτωση θα έχουμε για τις ε, θέσεις απασχόλησης, για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις από τη χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικό δηλαδή, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό. Πρόσφατα, οι υπηρεσίες μας δημοσίευσαν και μοίρασαν στην Επιτροπή Ρέτζι ένα φυλάδιο με τίτλο «Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία που συνεργάζονται για θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη». Το φυλάδιο έδινε πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων συνεργειών και τόνιζε ποιες πρωτοβουλίες είχαν ε, ψηλό δυναμικό. Παραδείγματο χάρη το επιτυχιακό πρόγραμμα της Ρουμανίας για την ανταγωνιστικότητα ή τα προγράμματα ε, καινοτομία στην ε, Βεσφαλία ή το εργαστήριο νανοτεχνολογίας Πορτογαλίας και Ισπανίας ή στην Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία άλλα προγράμματα ή ε, το πρόγραμμα Bonus στην Βαλτική. Μια άλλη ε, έμπρακτη απόδειξη των συνεργειών είναι ένα νέο επιτυχές εργαλείο που είναι η σφραγίδα αριστείας. Είναι ένα τίτλος ποιότητας που δίδεται σε προγράμματα τα οποία υποβάλλονται στο SME και στον ορίζοντα 2000 που καταφέρουν να επιτύχουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον αξιολόγηση, αλλά που δυστυχώ δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με βάση τον υπάρχοντα προπολογισμό. Αυτά τα πολύ ποιοτικά προγράμματα μπορούν συνεχεία να ψάξουν να βρουν εναλλακτική χρηματοδότηση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Και από τη στιγμή που δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία τον Νοέμβριο, όλε αυτέ οι προσδοκίε ε, υλοποιήθηκαν. Υπογράψαμε η Κορίνα Κρέτσου και εγώ πάνω από 3.200 τέτοιες φραγίδες αριστείας. Από όλα τα κρατημέλη. Προγράμματα δηλαδή από όλα τα κρατημέλη. Και παράλληλα έχουμε πάνω από 100 αρχές χρηματοδότησης που εκπροσωπούν και την πλευρά της έρευνας και της συνοχής, ούτως ώστε να κινητοποιηθούμε και να συνεργαστούμε για να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μέτρα για να υποστηρίξουμε την πρόταση γύρω από το, τη σφραγίδα αριστείας. Να συνημερώσω λοιπόν ότι συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες και το κάναμε για να μην υπάρξουν διαφορές ανάμεσα στις σφραγίδες ε, αριστείας και τους κανόνες ε, κρατικών ισχύσεων που πλέον δεν υπάρχουν αυτές, ε, αυτά τα προβλήματα για να μην υπάρχουν και σημεία ας πούμε έτσι που δημιουργούνται κόμματα, συμφόρηση κτλ. Η Κομισιόν δημιούργησε μια πλατφόρμα για να διευκολύνει την ανταλλαγή ε, πρακτικών και για να εντοπίσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα πιθανά εμπόδια για να εφαρμόσουμε απρόσκοπτα το, τη σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή αριστείας πιστεύω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2016. Και μάλιστα ήταν αναπάντηχη αυτή η επιτυχία. Το ερώτημα είναι, τελειώσαμε ή πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Όχι, δεν τελειώσαμε. Οι συνέργειες είναι σε μια διαδικασία πλούστευσης, αν θέλετε. Είναι μια δουλειά που δεν έχει τέλος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να προσπαθούμε όλο και περισσότερο και πιο διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα βελτιώσουμε και θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνέργειες, παράδειγμα χάρη το, της φραγίδα σε άλλους τομείς του ορίζοντα 2020, ε, η δράση ας πούμε, του Μαρή Κιουρί κτλ. Και, και στο μέλλον θέλουμε να εμπλέξουμε και τα JTI για να διερευνήσουμε περισσότερες συνέργειες με βάση τη θαυμάσια δουλειά που έχουμε ήδη κάνει στα πλαίσια των καθαρών ουρανών ούτως ώστε να βελτικοποιήσουμε την επίπτωση αυτών των προγραμμάτων μέσω συγκεκριμένων συνεργειών, ούτως ώστε να προχωρήσουμε πιο πολύ στην αεροναυπηγική. Νομίζω ότι από αυτή την έννοια ε, το Clean Sky, η καθαρή ουρανή, είναι ένα μοντέλο που πρέπει να το ακολουθήσουμε και σε άλλους τομείς. Ας αγγίξω τώρα ε, θέματα που θα σας παρουσίασει κανονικά η Επίτροπος Κρέτσου. Να ξεκινήσω με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης οι στρατηγικέ έξυπνη εξειδίκευση. Αυτέ οι στρατηγικέ έπρεπε από την αρχή να ε, ε, συνδυάζουν διάφορες χρηματοδοτήσεις και πρωτοβουλίε του ορίζοντα 2020, ούτως ώστε να συμπεριλάβουν και τους φορείς, οι οποίοι με τον ορίζοντα 2020 και με τη διαχείριση σε, στα, στην, στα πλαίσια της άλλων προσπαθειών ε, διαμορφώνουν τις στρατηγικές ε, έρευνας για την έξυπνη εξειδίκευση. Η Κομισιόν βοηθάει συνεχώς τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για να αναπτύξουν τις ε, στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης κυρίως μέσω των πλατφόρμων που έχουν δημιουργηθεί, τις πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στη Σεβίλη στην Ισπανία με τριπλό σκοπό. Να επιταχύνουμε την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών έξυπνης εξειδίκευση να διευκολύνουμε την διεθνική συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και τρίτον, να δημιουργήσουμε μία σειρά από θεματικές έξυπνες εξειδικεύσεις ε, και σχετικές πλατφόρμες. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις τέτοιες πλατφόρμες, μία για την ενέργεια και την ενεργειακή καινοτομία, μία δεύτερη για, την, ε, για το βιομηχανικό εξυγχρονισμό και μία τρίτη για τα, τη γεωργία και τα τρόφιμα. Αυτές οι πλατφόρμες και άλλες πλατφόρμες στο μέλλον θα μας βοηθήσουν τόσο ώστε να έχουμε αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων των διαφορετικών ταμείων και να υπάρξει και μόχλευση με επιπλέον πόρους από τον ορίζοντα 2020, αλλά και ιδιωτική χρηματοδότηση από το ΕΦΣΙ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή η προσέγγιση με τις πλατφόρμες ε, είναι η συνέχεια ενός καλού προγράμματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας που μας ε, επέτρεψε η συνεργασία από, μεταξύ 30 περιφερειακών κυβερνήσεων να περάσει σε συγκεκριμένες αλυσίδες αξιών, ούτως ώστε να περάσουμε σε επαφή με τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές και τα ερευνητικά κέντρα. Επίσης υπάρχει μια εταιρική σχέση για επενδύσεις στην έξυπνη εξειδίκευση για να υποστηριχθούν αυτέ οι πλατφόρμες και να υπάρξει εξυγχρονισμό, ούτω ώστε να υπάρξει πραγματική συμμετοχή από τι επιχειρήσει. Και τέλο, ε, δύο λόγια για τη σκάλα αριστεία. Η πρωτοβουλία που έχει, ξεκίνησε εδώ στο Κοινοβούλιο με ένα πιλωτικό πρόγραμμα που εντοπίζει ε, συνέργειες ε, σε 13 κράτη-μέλη την ανάγκη να γίνει μια διαδικασία αέναη που θα εμπλέκει τις επιχειρήσεις, τη ερευνητικά κέντρα και την ε, εκμετάλλευση της ε, διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας. Ε, έχουμε 11 εθνικές εκδηλώσεις που έχουν ήδη λάβει η χώρα. Αυτό το project θα διευρυνθεί και στα αλλα κρατημέλη, κράτη-μέλη, πέρα τα 13 δηλαδή, ούτως ώστε να εμβαθύνουμε και εκεί τις συνέργειες. Ο Στίβεν Κόφι είπε ότι οι συνέργειες είναι η βελτίωση του δικού μου ή του δικού σου τρόπου. Γιατί είναι ο δικός μας τρόπος. Σας ευχαριστώ και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε Επιτρόπε και πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Έλλερ. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι ε, θα υπερβούμε πραγματικά τον χρόνο που προβλέπετε για την ε, σημερινή ολομέλεια. Θα φτάσουμε μέχρι και 11.20 όπω έχουν τα πράγματα. Δεν θα δεχτώ μπλε κάρτε, αλλά θα δεχτώ ε, catch the eye. Ο κύριο Έλερ για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι ότι με τις σημερινές συζητήσει για το κοινό ψήφισμα για τις συνεργίες μεταξύ των θετικών ταμείων και του προγράμματος ορίζοντας 2020 ε, θέτουμε ένα ορόσημο. Ξεκινάμε τη συζήτηση ουσιαστικά για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικά και μία απάντηση για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για τον πολίτη, τι μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει η Ευρώπη για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη. Η σημερινή λοιπόν συζήτηση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εκκίνηση. Δεν αποτελεί μία τεχνική συζήτηση για τον προπολογισμό. Η καινοτομία είναι ουσιώδου σημασία για την κοινωνική ανάπτυξη, για την οικονομία, για την πρόοδο της Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κοινοτομίας έχουμε κάνει περικοπές. Έχουμε θέσει άλλα σημεία επικέντρωσης και το έχουμε πληρώσει πικρά αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι σημαντική. Είναι σημαντική για να κατανοήσουμε ότι κάποια προβλήματα για την κατανομή, για παράδειγμα, των πόρων για την καινοτομία, δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε αν δεν θέσουμε επί της αρχής κάποια διαστατικά ζητήματα, τα διαστατικά ταμεία, αν δεν μεταρρυθμιστούν. Προκειμένου οι αριστούχοι επιστήμονες να έχουν διαστατικά τα μέσα για να μπορούν να προχωρήσουν. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι βασική η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ευχαριστώ η κυρία Καμπεσόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το να πετύχουμε το στόχο του 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 οικονομικός πώς είναι εφικτό. Πάνω από 120 εκατομμύρια ε, από τα ταμεία. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε όλους τους στόχους ε, πώς θα λειτουργήσουν τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένες καλές πρακτικές. Αν τις ξέρουμε να τις μάθουμε κι εμείς. Επίσης μπορούμε να ξέρουμε αν μπορούν, μπορεί η νομοθεσία να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε δυσκολία. Νομίζω επίσης ότι είναι ε, σημαντικό να διευκολύνουμε τη διασύνδεση ανάμεσα ε, στα θεσμικά όργανα με τα προγράμματα έξυπνων στρατηγικών τα οποία αναπτύσσονται για αυτές τις ε, προτεραιότητες που ανέφερε η Κομισιόν με την ε, έρευνα ε, και με ιδιωτικά και με δημόσια ερευνητικά κέντρα. νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση με όλα αυτά τα πράγματα που θα τα εξηγεί πολύ ξεκάθαρα. Κύριε Τόμασιτς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Το ECR υποστηρίζει την συνέργεια ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και τον ορίζοντα 2020 με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο ορίζοντας 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την καινοτομία και την αριστεία στην επιστήμη, για την ε, τις μεταλλαγές που πρέπει να επέλθουν ε, για να προσαρμοστεί η επιστήμη και να, γίνει πιο, ε, να είναι πιο ανθεκτικά τα αποτελέσματα ε, της έρευνας ως προς τις μελλοντικές ε, προκλήσεις. Ε, το, η ευθυγράμμιση προς το σχέδιο Juncker δεν είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι αν συνεχιστεί, α, συνεχίσουμε σε αυτή την άγουσα θα υπονομεύσουμε την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα του ορίζοντα 2020. Είναι ξεκάθαρες οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αριστεία στην επιστήμη για την ε, οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει αυτό να έχει επιρροχή σε σχέση με ε, σαθρά μεγαλεπίβολα πολιτικά σχέδια η πολιτική συνοχή σε αυτή την προγραμματική περίοδο δεν θα πρέπει να συνδεθεί με τον ορίζοντα 2020 γιατί διακινδυνεύουμε μια πολύ σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Φαν Μίλτον, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύει σε κοινοτομία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό οδηγεί σε ανέσταση, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Αλλά το γεγονό είναι ότι έχει μείνει πίσω η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό τι σημαίνει ότι κάθε ευρώ που ταπανάτε στον κοινοτικό προβολογισμό πρέπει να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό ήταν και το μήνυμα τη Επιτροπή Juncker όταν ε, ανέλαβε τα καθήκοντά τη. Μα υποσχέθηκε πέρσι ότι θα είναι μεγάλο ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά τι επενδύσει ε, στην καινοτομία. Και η Επίτροπος Κρέτσου μας ανακοίνωσε την ε, ε, Seal of Excellence τη φραγίδα αριστείας. Δυστυχώ τα πράγματα θεωρώ ότι παραέμειναν σε επίπεδο δεσμεύσεων και υποσχέσεων. Και στην πράξη βλέπουμε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ιδιαίτερα αυτές οι υποσχέσεις σε ό,τι αφορά την απόδοση. Οι επιχειρήσεις ε, στα χαρτιά έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά η υλοποίηση στην πραγματικότητα, στην πράξη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και έτσι λοιπόν ο ορίζοντας 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα ταμεία για να υπάρξει αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να απλοποιηθούν αυτά τα μέτρα και αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να προδιαγράφονται μόνο από τις Βρυξέλλες, από κάποιο γραφείο. Θα πρέπει να υλοποιούνται με τη βοήθεια ε, εμπειρογνωμόνων. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, πιο κοντά στη βάση. Οι συνέργειες λοιπόν θα πρέπει να έχουν πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό, να επενδύσουμε και να υπάρξει ανάπτυξη και θέση εργασία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό και σομαζέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Εδώ και πολύ καιρό ζητούμε ε, τη ε, συνέργεια ανάμεσα στον τα 2020 και τα διαρθρωτικά ταμεία. Προσοχή όμως, οι αρχές ε, της συνοχής θα πρέπει να διαφυλαχθούν και οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες παραδείγματος χάρη, δεν θα πρέπει να στερηθούν ε, τα ωφέλη του ορίζοντα 2020. Επίσης θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί ε, τόσα πολλά μικρά προγράμματα, τόσες ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020. Ε, ενδεχομένως ε, φανταζόμαστε είναι υπερβολικά μεγάλα τα προγράμματα, ενδεχομένως είναι εξαιρετικά περίπλοκη η διαδικασία και νομίζω για αυτό το λόγο ταυτόχρονα με τη συνέργεια θα πρέπει να προωθήσουμε την απλούστευση και αναμένουμε τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας που συγκρότησε για αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαραγκάλη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Χαιρόμαστε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε να βρείτε τις, ε, αυτές τις συνέργειες. Έχουμε την συνοχή στον προπολογισμό ε, και έχουμε και τα διαφορετικά ταμεία. Έχουμε τα ερευνητικά προγράμματα που αναζητούν την αριστεία. Έχουμε την πολιτική συνοχή όμως που συχνά αλλάζει και προσπαθεί να ρυθμίσει κοινωνικά και πραγματικά προβλήματα, αλλά με ελάχιστους πόρους. Είδαμε τι γίνεται, ότι μερικές φορές τα αεροδρόμια είναι ε, γεμάτα κόσμο και άλλα αεροδρόμια είναι άδεια. Η Κομισιόν θέλει να βοηθήσει στη συνεργασία, στη συνέργεια με διάφορα προγράμματα, όπως παραδείγματο χάρη το, με το πιλωτικό πρόγραμμα που προωθήσαμε για την οικονομική συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Είναι σε φάση εκτέλεσης, αλλά πρέπει να ξεχνάμε τι κρύβεται πίσω από αυτήν την πολιτική. Δεν θα πρέπει να αναλάβουμε στόχους που δεν αρμόζουν στις διάφορες πολιτικές. Ούτε επίσης λόγω της συνέργειας θα πρέπει να κάνουμε πορεία προς τα πίσω. Έχουμε θετική άποψη για τις εξηγήσεις σας. Μας αρέσει αυτή η σφραγίδα αριστείας, αλλά προσοχή, θα πρέπει να μην κάνουμε μόνο ε, προσπάθειες marketing, θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των ε, περιφερειών ε, και των κρατών. Κύριε Μαραγάλη, μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούσα να παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ο κύριος Νταμάτο, 1,5 λεπτό. Ή κυρία Νταμάτο. Η συνέργεια μεταξύ του ορίζοντα 2020 και διαφορετικών ταμείων μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε τα διευθυντικά ταμεία θέλουν να οικοδομήσουν το απαραίτητο δυναμικό ε, με βάση τις ανάγκες των περιφερειών που έχουν περισσότερα προβλήματα. Με μια διαχείριση και περιφερειακή και εθνική. Ε, το ορίζοντα σε 2000 ε, προωθεί την αριστεία. Τα διευθυντικά ταμεία αφορούν μία περιφέρεια και μία περιφέρεια στηρίζεται μέσα σε μία ε, εφταετία, ενώ τα, η χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020 γίνεται με βάση τα κριτήρια του ανταγωνισμού. Επομένω, είναι διαφορετική η χρηματοδότηση. Στην πράξη, οι συνέργειε έχουν νόημα για να βρούμε ε, του πόρου που δεν χρησιμοποιούνται σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα αξ, ε, αριστείας το οποίο δεν κατάφερε να χρηματοδοτηθεί από αλλού. Αλλά η υποκρισία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Από τη μία, μα καλεί να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία και από την άλλη, ε, βγάζει 22,2 εκατομμύρια από το Horizon για να τα δώσει στο σχέδιο ε, Juncker που είναι αμφίβολης χρησιμότητας και μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση με, τις, ε, με τους στόχους πολιτικής συνοχής. Επομένως, πηγαίνουν προς μια επικίνδυνη κατεύθυνση, προς μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, όλο και περισσότερο. Μια, ένα ρήγμα όλο και περισσότερο, ανάμεσα σε κράτη πιο ανεπτυγμένα και λιγότερο ανεπτυγμένα μην σα κάνει εντύπωση που βλέπουμε την αντίδραση των λαών αντίον τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ε, παρετούμαστε από την ίδια της την ιδέα τη Ευρώπη. Ο κ. Λερόι για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά παραδείγματα που μα δώσατε. Αλλά τα πράγματα πρέπει και μπορούν να βελτιωθούν σε ό,τι αφορά τις συνεργίες μεταξύ ορίζοντα 2020 και άλλων μέσων και εργαλείων. 90% των επενδύσεων στον ορίζοντα 2020 καταλήγει στα παλαιά κράτη-μέλη. 80% των διερθωτικών ταμείων πάει στα καινούρια κράτη-μέλη. Είναι δύο σημαντικά λοιπόν ταμεία ξεχωριστά και απαραίτητα. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Δεν είναι καλό λοιπόν αυτό. να υπάρχει κάπου πλούτο και κάπου άλλο τελμάτο, Γιατί η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την καλή και ισορροπή ανάπτυξη, την καλή ε, και ενταφική συνοχή. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ε, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μία να υπάρχει το συντηρητή του Λονδίνου και από την άλλη να υπάρχει και η πετρόση η οποία υστερεί. Έτσι λοιπόν οι πολίτες αποστρέφονται την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση, ζητάμε λοιπόν ένα καινούριο συνδυασμό που θα βασίζεται στην καινοτομία και ενίσχυση των προϊόντων και των υπηρεσιών που βασίζονται στην καινοτομία. Αυτό είναι δυνατό λοιπόν. Έχουμε λοιπόν 60 δισεκατομμύρια για την καινοτομία, για την έξυπνη, ευφύ εξειδικευσή. Ο Ρόμπερτ Μάντελιν ε, αυτή την εβδομάδα ανέφερε την αποστολή του για την ε, καινοτομία, ένα σύμφωνο καινοτομία με ένα νέο τρόπο για την συνεργασία. Το δικό μας ψήφισμα και η δική σας ιδέα για την ευρωπαϊκή καινοτομία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ επίκαιρα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή αυτή που θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι δεν επιτρέπονται μπλε κάρτε σήμερα το βράδυ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σα ευχαριστώ για την κατανόησή σα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοτζολίνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είναι σαφέ ότι συζητάμε για μια πολιτική που λειτουργεί σήμερα, δρά σήμερα και με του ισχύοντε πόρου. Μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων που έχουν προγραμματιστεί ε, για τις περιφέρειες ε, φτάνουμε στα 100 εκατομμύρια επενδύσεις και 80 εκατομμύρια από τον ορίζοντα 2020. Μιλάμε δηλαδή για ένα σημαντικό πακέτο πόρων που τα έχουμε για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, για να δρομολογήσουμε ξανά την καινοτομία, για τις επιχειρήσεις μας, για τα ερευνητικά μας κέντρα και για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις, κυρίως αυτές των νέων. Το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καλό θα ήταν λοιπόν να το ελέγξουμε το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε πολύ προσεκτικά τα επόμενα χρόνια για το πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο ταμεία και να γράψουμε τις σελίδε του μέλλοντος, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμπληρωματικότητα, μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο ταμεία. Φερρυπίν, να εξασφαλίσουμε όπως κάνετε μέρη στην Επιτροπή, ότι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν ε, τους περιφερειακούς πόρους από τα διευθυντικά ταμεία, να χρηματοδοτηθούν από αλλού. Ένα λεπτό. Ο κ. Καράσνοντοψκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η συνέργεια ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και στα διαφορετικά ταμεία έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σε κάποια κράτη-μέλη ότι θα πετύχουν την επιστημονική αριστεία χρησιμοποιώντας αυτά τα ταμεία. Αυτός ο στόχος όμως δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει υλοποιηθεί. Και το ρήγμα ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη μεγαλώνει. 13 νέα κράτη-μέλη έχουν πάρει μόνο το 5% του συνολικού προϋπολογισμού υπό τον ορίζοντα 2020. Αν θέλουμε πραγματική συνέργεια θα πρέπει να δράσουμε και σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί υιοθετεί του κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει, για του ελέγχου και τι διαδικασίε. Το ποσοστό στη χρηματοδότηση είναι διαφορετικό ανάλογα με το, ανάλογα το αν πρόκειται για τα διαφορετικά ταμεία για τον ορίζοντα 2020. Υπάρχουν και άλλε διαφορέ. Ανάλογα με τη γλώσσα των αιτήσεων. Το αυτή η σφραγίδα αριστεία δεν είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προσαρμόσει τι διαδικασίες. Η διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά, γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία και στον ορίζοντα 2020. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Κυρία Βέρινγκ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, Αγαπητοί Επιτροπέ, αγαπητοί συναδελφοί, το ψήφισμα που έχουμε επιτάπητος είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα. Πρόκειται για μια ευκαιρία τέτοια υλοποίηση των συνεργειών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το τρέχον κείμενο δεν αναφέρεται μάλλον δεν επηρεάζει το κείμενο των δύο προγραμμάτων, αλλά τονίζει το θέμα της συμπληρωματικότητα, Το ορίζοντα 2020 θέτει το κριτήριο τη αριστείας, αλλά το προπολογισμό δεν επαρκεί για να υποστηριχθούν όλα αυτά τα πολλά υποσχόμενα προγράμματα. Αυτή η σφραγίδα αριστείας φροντίζει προκειμένου τα θετικά ταμεία να μπορούν να εντοπίζονται το, το συντομότερο δυνατόν και να υποστηρίζονται λόγο. Αυτό είναι καλό παράδειγμα για τη συνέργεια αυτή και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιούν αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια ευκαιρία να τονίσουμε και να τονώσουμε την επιστήμη και την καινοτομία και να δώσουμε μια εξασφάλιση για τις θέσεις απασχόλησης στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έθριτς δεν είναι στην αίθουσα και άρα το λόγο παίρνει κατευθείαν ο κύριος Μπούζεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Ναι, ε, κάνουμε τώρα την ενδιάμεση αναθεώρηση του ορίζοντα 2020. Έχουμε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, έρευνα. Και τώρα βλέπουμε στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 πώς γίνεται η κατανομή των πόρων και για τα διαρθρωτικά ταμεία το ίδιο. Όλος ιδιαίτερος όμως μας απασχολούν οι διαφορές ανάμεσα στα 13 νέα κράτη-μέλη και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τους πόρου αυτού των διαστατικών ταμείων να τους χρησιμοποιούμε πραγματικά για μελλοντικέ επενδύσεις και χρειαζόμαστε και την ολοκλήρωση του ε, προγράμματος ε, πλαίσιο αλλά και την ε, εφαρμογή του ορίζοντα 2020. Αυτή η συνέργεια διαρθρωτικών ταμείων και ορίζοντα 2020 είναι πολυδιάστατη. Όμως η ευφυής εξειδίκευση, παραδείγματο χάρη, ε, δεν ταιριάζει παρά μόνο με τα κριτήρια των διαρθρωτικών δαμείων και όχι με τον ορίζοντα 2020. Αυτή η σφραγίδα αριστείας δεν έχει λειτουργήσει τόσο καλά όσο νομίζαμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ομοιόμορφα πρότυπα που θα ισχύουν ε, διατομιακά για όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε Ε, επιστήμονες ε, από τα νέα 13 κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε επιστημονικά δίκτυα και σε ε, ομάδες εργασίας επιστημονικών συμβούλων. Ευχαριστώ. Κύριε Τόια, συμφωνούμε, Επίτροπε, με αυτά που είπατε και με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Καινοτομία. Και όλοι ξέρουμε ότι σήμερα οι λέξεις κλειδιά για μια αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως σε μια τόσο στρατηγική πλευρά όπως η έρευνα και η πολιτική συνοχής είναι συνέργεια, συμπληρωματικότητα, συγκέντρωση θεματική ε, σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Για όλα αυτά τα θέματα, συνδυαστικά, ας το πούμε έτσι, που μας επιτρέπουν την χρήση για το ίδιο πρόγραμμα ε, διαφορετικών ταμείων και προγραμμάτων και κονδυλίων, ε, που θα, χάρη σε εμάς θα συγκλίνουν για να μας επιτρέψουν να, φτιάξουμε, να έχουμε κατλά αποτελέσματα για την ψηφιοποίηση, για την ε, βιομηχανική έρευνα, για την ανταγωνιστικότητα, για την αξιοποίηση των τεχνολογικών ανακαλύψεων κτλ. Όπως είπε και η κυρία Καμπεθόν Ρούις, όλες αυτές ε, οι νέες, ε, όλοι αυτοί οι νέοι τομείς πάνω σε αυτούς δεν υπάρχει ε, αρκετή γνώση. Δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις συνέργειες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια, να, γίνουν γνωστές οι, βέλτιστες πρακτικές και να βοηθήσετε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Μιχαήλωβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, συζητούσαμε τα προβλήματα της ε, συνέργειες ανάμεσα στα διευθυντικά ταμεία και τον ορίζοντα 2020 μας απασχόλησε ο συντονισμός των διάφορων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συζήτηση δείχνει ότι είναι κοινή ανάγκη ε, να επιτύχουμε μεγαλύτερες επενδύσεις ε, για να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργία και δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στο, επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να μας αποσχολήσει είναι η εφαρμογή, επιτόπια εφαρμογή. και η συνεργασία ανάμεσα σε διάφορα προγράμματα. Έχουμε ε, στόχους κοινού, όπως ε, η τόνωση της ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κοινού μας στόχους. Ευχαριστούμε για κάρτα, αλλά ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Επιτροπή δίνει θεωρητικούς προς προσανατολισμούς για να υπάρξουν οι συνέργειες μεταξύ των διαθωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων και του ορίζοντα 2020 δεν έχουμε τόσα πολλά λεφτά, αλλά η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ε, χρήζει όχι ποιότητα, ε, ποσότητας, αλλά καλή διαχείριση για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και να ε, καταρρύψουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια. Επίσης πρέπει να υπάρξει έξυπνη εξειδίκευση με προγράμματα διαφορετικά ε, στα πλαίσια του, του ίδιου πλαισίου ή παράλληλα προγράμματα. Επίσης θα πρέπει να επιλύσουμε προβλήματα για να προωθήσουμε τη συνέργεια αυτά που σχηματοδοτούν τα διεθνωτικά ταμεία σε εθνικό επίπεδο θεωρούνται κρατικέ ενισχύσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Όταν μιλάμε για φορεί που, που έχουν οικονομικέ δραστηριότητε και τέτοιου τύπου που δεν του επιτρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον ορίζοντα 2020. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να υλοποιήσουμε τους στόχους μα. Αυτή η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερε καινοτόμε μικρομεσαίε επιχειρήσει για να φτιάξει ε, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο η Βρυξέλλες ή το Βερολίνο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και τα Κανάρια και η Μούρθια ε, που παράγουν τρόφιμα ή ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο θα, υπάρξει θέσεις, θα υπάρξουν θέσεις απασχόλησης. Επομένως πρέπει να δούμε τις δραστηριότητε όλων των οικονομικών φορέων. Θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να είναι σίγουροι ότι δεν σπαταλάμε ούτε ένα ευρώ λόγω γραφειοκρατίας και λόγω επικαλύψεων. Και οι συνέργειες είναι ο καλύτερος ε, σύμμαχός μας για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Κουστινάρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε. Να σας ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι αναφέρατε στο πρόγραμμα Γιατί πρόκειται για μια επιτυχία για τις συνεργίες μεταξύ των ευρωτικών Ταμείων και του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Πραγματικά θαύματα ε, πετυχαίνουμε. Το πρόγραμμα Light λοιπόν ε, ε, αναπτύσσεται στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά αφορά μεγάλη έρευνα και γενοτομία από όλο τον κόσμο. Αυτό θα μεταβάλει την ε, Ευρώπη σε μεγάλη δύναμη σε ό,τι αφορά τα πρόγραμματα laser. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό στη Ρουμανία θα απασχολήσει 600 επιστήμονες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από όλο τον κόσμο και θα έχει επιπτώσεις και επιδράσεις ανάλογες με αυτές του ΣΕΡΝ. Γι' αυτό λοιπόν καθλωσορίζω τις συνέργειες και είναι καλό να μιλάμε για τη χώρα μου και τις συνέργειες γιατί αποτελούν αυτό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και τώρα για ένα μισή λεπτό το λόγο και ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρα, κυρία Μακίνας. Συνεργάζεστε μαζί μας και στην Επιτροπή Στούα και για μας στην Επιτροπή ΣΤΟΑ. Πώς μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε στην έρευνα και στην κινητομία στη, στα spin-off, ε, σε θέματα μ, τέτοιων προγραμμάτων. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να επενδύσει προς την κατεύθυνση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ο ορίζοντα 2020 και τα τελευταία ταμεία αποτελούν ένα υπέροχο παζλ και παρέχουν το σωστό πλαίσιο για όσους θέλουν να σημειώσουν αποτελέσματα και να, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πλούτο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να είναι αυτοαπασχολούμενοι για να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην στον του 2020 και γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε και την ευφυή εξειδίκευση. Θα πρέπει να είναι σαφές το πώς αυτές οι νέες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν στο σωστό τομέα και η κατάρτιση και η εκπαίδευση λοιπόν θα παίξουν ρόλο κλειδί. Και Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, υπόλυβα, να υποβάλει προτάσει προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή Μόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα λεπτό, η κυρία Κόμπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επιστήμη είναι το μέλλον και οι, οι κορυφαίοι επιστήμονες θα πρέπει να συνεργάζονται στους διάφορους τομείς. Αυτή η κοινοτομία είναι που δίνει πνοή στην οικονομία και έτσι μακροπρόθεσμα αυξάνει την ανταγωνιστικότητά μας. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 βοηθάει την Ευρώπη να αναπτυχθεί προς μία πιο ευφύ κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε έρευνα στους τομείς αυτού στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτροπό για το περιφερειακό πρόγραμμα πόνους. και τα κρατημέλη και η Ένωση δεν μπορούν να περικόπτουν πόρους στο μέλλον, για το μέλλον. Ο ορίζοντας 2020 θα πρέπει να έχει σωστή ποιότητα και σωστό επίπεδο. Γιατί έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη να πετύχει την ανταγωνιστικότητα και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ισορροπία και ομοιογένεια μεταξύ των περιφερειών και τώρα πιστεύουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια χώρα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή έρευνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή με την με Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ και ένα λεπτό κύριο Μπόκοβιτ. Ευχαριστώ. Συζητήσαμε ήδη Πρωτοβουλία για τους νέους. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας παρουσίασε τα αποτελέσματα του ΕΦΣΙ και τώρα συζητάμε τον ορίζοντα 2020 και τα διαρθρωτικά ταμεία. Όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να την εκρίζωση τις στόχους, δηλαδή από τη μία πλευρά και από την άλλη. Προσπαθούμε να βρούμε νέες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η ευφυής e εξειδίκευση καθιερώνεται όπως και ορίζοντας 2020. Όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα και διαπιστώνουμε πως τα νέα κράτη-μέλη απορροφούν 95% των κονδυλίων, είναι ξεκάθαρο ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να βρει ένα σύστημα ότως ώστε ε, να μπορέσουν να υποφεληθούν τα νέα κράτη-μέλη και από τον του 2020 και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα ανακύψουν και άλλες, ε, άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ η κυρία Ροντρίγκε, Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, έχουμε τις διάφορες συνέργειες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές επενδύσεις και τις εθνικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας. Χρειαζόμαστε πολιτική συνοχή για τις επιμέρους περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωση. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, ε, γιατί τιμωρούνται έτσι τα κράτη-μέλη για την πρόσβαση στα κονδύλια των διορθωτικών ταμείων. Ε, πώς ε, εννοείται την πολιτική σύνοχη, την αποφασίζει το είναι πώς γίνεται με την λιτότητα που έχει επιβάλει η Τρόικα τα τελευταία τέσσερα χρόνια να τιμωρείται η χώρα ε, γιατί ε, ε, το 2015 κατά 0,14% δεν τήρησε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Τιμωρείται η χώρα μας διότι δεν ακολουθεί αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ε, επίτροπε, ε, εσείς και οι συνάδελφοί σας ξέρετε πολύ καλό ότι αυτή είναι η κατάσταση, τιμωρείται η χώρα και το ξέρουν οι αγορές, το ξέρει και ε, το ΕΚΟΦΗ. Thank you for one minute, Mr. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Λεβαντόσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνέργεια, καταπληκτική λέξη σημαίνει ότι οι προσπάθειες και μέσα ε, συνδυάζονται αντί να υπάρχει κατακαιρματισμός των προσπαθειών. Δεν υπάρχει ενιαία απορρόφηση των μέσων ε, ε, και ε, ε, ομοιόμορφη κατανομή των κονδυλίων στο Νότο και στα νέα που δεν είναι και τόσο νέα χρησιμοποιούν τα τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων ενώ τα παλιά κράτη-μέλη τον τίτλο 1α. Εγώ νομίζω πως Όντω θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ερευνητικά προγράμματα, όμω θα πρέπει να ξέρουμε ότι ε, ακαδημαϊκοί φορεί δεν συνεργάζονται επαρκώ με την επιστημονική κοινότητα και χρειαζόμαστε καλύτερα μέσα, χρειαζόμαστε διαδοτικά τμήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μέρη της, κυρίως αυτές τις, ε, τα νέα παλιά κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Κύριος Μπούντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ να βρει μηχανισμούς και μοχλούς για να εκφράσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και για να μειώσει ταυτόχρονα τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική συνοχή εν το συνόλο της αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους που είναι πολύ σημαντική προφανώ. Πέρα από την ευελιξία, πέρα από τι νέε πραγματικότητε στις οποίε πρέπει να προσαρμοστούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνέργειε μεταξύ των πέντε διαφορετικών ταμείων, αλλά και μεταξύ άλλων σημαντικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα και τελικά να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση. Η απλούστευση επίσης ή σαφείς κανόνες για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων και η διαφάνεια θα πρέπει να είναι προτεραιότητες για την Κομισιόν. Όλα αυτά θα πρέπει να μας δώσουν εγγύηση ότι τα ταμεία θα είναι προσπελάσιμα από όλα τα κράτη-μέλη ε, επίσης όρις. Και τώρα πάμε στο, στη διαδικασία Catch the Ο κύριος ε, Μουράγιας είναι ο πρώτος ομιλητή. Μαριά, συγγνώμη. Ορίζοντας 2020 υποστηρίζει τη στρατηγική ευρώπη 2020 και έχει σαν στόχο να ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη της ένωσης. η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 16 δις ευρώ για το διάστημα 2016 2017 που περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας με χρηματοδότηση 1 δις ευρώ καθώς και την κυκλική οικονομία με 670 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση παράλληλα μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών η αναθεώρηση των κρατικών επιδοτήσεων και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. δεδομένη ωστόσο τη υψηλή ανεργία που παρατηρείται σε ορισμένα κράτη μέλη τη ένωση και ιδίω στην ελλάδα υπάρχει ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την καινοτομία την έρευνα και την ανάπτυξη καθώ και ανάγκη για αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Ιακοβτσίτς. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνεργίες χωρίς αμφιβολία είναι μια πάρα πολύ όμορφη λέξη και την χρησιμοποιώ συχνά στις πολιτικές μου ομιλίες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Προφανώς και χρηματοδοτείται ορίζοντας 2020 και τα ποσά αυτά τα βλέπουμε και στα διαφορετικά ταμεία και στην πολιτική συνοχή. Και γι' αυτό λοιπόν θα συστήνω προσοχή, λαμβάνοντα υπόψη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αν πάρουμε και ένα τμήμα του προγράμματος του Juncker για να υποστηρίξουμε πολλά από τα σημαντικά προγράμματα τα οποία ε, μέσω των ε, διαθετικών ταμείων ε, χρηματοδοτούνται και είναι πολύ σημαντικά για τις υποδομές στα νέα κράτη-μέλη. Ας βρούμε λοιπόν μια ε, δημιουργική, ένα δημιουργικό τύπο και να υπάρξουν λοιπόν συνεργίες μεταξύ όλων των μέσων και όχι μόνο μεταξύ αυτών των δύο γιατί αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες εκεί που υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ήρθε η Επιτροπή εδώ να μα μιλήσει για τι συνέργειε ανάμεσα στα διευθυντικά ταμεία και τον ορίζοντα 2020. Η ίδια η Επιτροπή που στο πρόγραμμά τη έχει εφαρμογή απαράδεκτων δικαιολόγητων κυρώσεων κατά τη Πορτογαλία που παραβιάζουν τον κανονισμό ε, των διαρθρωτικών ταμείων. Η Πορτογαλία ε, συνέβαλε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ξεκάθαρα και ε, δηλαδή στο πρόγραμμα που υπήρχε πριν από τον ορίζοντα 2020 και που ε, χρωματοδοτούσε την έρευνα για τους πλούσιους που τώρα ζητάνε να επιβληθούν επικυρώσεις κατά της Πορτογαλίας. Ε, θα πρέπει να το βάλετε στο κεφάλι σας ότι η Πορτογαλία θα επιβιώσει, η Πορτογαλία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα διορθωτικά ταμεία γιατί ε, τα λεφτά που παίρνουν από τα διευθυντικά ταμεία τα παίρνετε πίσω και με το παραπάνω, με τους στόχους ε, και είναι, ε, μη, είναι αθέμητες, είναι αδικαιολόγητες. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην Πορτογαλία είναι απαράδεκτο το, το μαρτύριο στο το οποίο έχετε επιβάλει στη, στο λαό της Πορτογαλίας. Ευχαριστούμε ο κύριος Νοβακόφ ένα λεπτό. Τι? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι χρειάζεται ενότητα ε, για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τον ορίζοντα 2020. Χρειάζεται ομοιομορφία προς τα πρότυπα. Μόνο έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τι εννοώ. 90 εκατομμύρια μέχρι το 2020 αυτός είναι ο προϋπολογισμός και ενισχύουμε ε, τη συνέργεια με τα διορθωτικά ταμεία και ο προϋπολογισμός εκείνη 350 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε ευέλικτα εργαλεία για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, την ε, μελλοντική έρευνα για τους Ευρωπαίους. Πώς μπορούμε να ε, ε, ε, περιμένουμε από τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τόσο περίπλοκα εργαλεία οι δικαιούχοι δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η διαδικασία. Χρειάζεται να συνδυάσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα και τα κεφάλαια που ε, προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρέπει να ε, συνδυάσουμε 500 διαφορετικά προγράμματα και σίγουρα πολλαπλασιαστούν τα καλά παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να μιμηθούμε. Ευχαριστούμε, Επίτροπος Μοέντας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λόγω τριών πραγμάτων. Πρώτον, λόγω του ότι όλοι συμφωνούμε για τη σημασία των συνεργειών, για να έχουμε καλύτερη επιστήμη και καλύτερη καινοτομία. Δεύτερον, συμφωνούμε ότι σε διάφορα έργα και προγράμματα και μέσα τα έχουμε καταφέρει. Τα παραδείγματα μιλούν από μόνα τους, είναι πολύ ευλώτα. Τρίτον, συμφωνούμε, παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, ότι είναι μια συνεχιζόμενη ομαδική προσπάθεια και πρέπει να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, διάφορες υπηρεσίες, οι λαοί, οι εθνικές κυβερνήσεις και δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε περισσότερες συνέργειες, να σκεφτούμε εφάνταστα, να δημιουργήσουμε νέα μέσα και εργαλεία που θα δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα. Έχετε λοιπόν την αμέριστη δέσμευσή μου και της Επιτρόπου Κρέτσου ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να δώσουμε περισσότερα τέτοια παραδείγματα όπως αυτά που ακούσατε σήμερα. Αλλά αυτό για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε βοήθειά σας. Χαίρομαι για την υποστήριξη, χαίρομαι για όλες τις ιδέες, για τις ερωτήσεις. Μείνετε ήσυχοι. Όλα τα σημεία τα οποία ακούσαμε σήμερα εδώ θα τα λάβουμε υπόψη μας στη δουλειά μας στον προβληματισμό μας και σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ιδέες. Δεν αποκλίνω τις δικές μας ιδέες. Νομίζω ότι δείχνουν πόσο προσιλωμένοι είμαστε προς τον κοινό μας στόχο όλοι. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση.